παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής εκδόσης εταιρείων στην Ευρώπη. Έχετε το λόγο κύριε Κόχ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, πώς θα φτάσει κανείς από τη Βαϊμάρη στη Λισαβόνα. Δεν είναι εύκολο ερώτημα αυτό. Οι ανάγκες των ταξιδιωτών ποικίλουν κατά πολύ άλλοι θέλουν να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, άλλοι θέλουν να ακολουθήσουν περισσότερο βιώσιμο τρόπο μεταφορών, άλλοι θέλουν ως τουρίστες να ψάξουν το δρόμο που θα τους οδηγήσει κοντά στα περιφέρεια. Αυτοί που θέλουν να επιλέξουν τη διαδρομή τους έχουν πολύ λίγες επιλογές. Δυστυχώς πολλές φορές οι προσφορές περιορίζονται μόνο ε, εντός των συνόρων μίας και μόνης χώρας και πολλοί προσφεύγουν στη μοναδική εναλλακτική λύση που είναι η χρήση του ιδιωτικού του επιβατικού αυτοκινήτου. Θα μπορούσαμε να έχουμε το όραμα της μεταφοράς από πόρτα σε πόρτα με ένα και μόνο εισιτήριο που θα συνδυάζει πολλά διαφορετικά είδη μεταφοράς πέρα από εθνικά σύνορα. Υπάρχουν πολλά εμπόδια και πολλές δυσκολίες για να υπάρξει ένα τέτοιο πολυτροπικό σύστημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με συστήματα πληροφόρησης, έκδοσης εισιτηρίων και ενημέρωσης του κοινού για τα δρομολόγια. Θέλουμε να έχουμε δίκαιη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες ε, για τις ε, διαδρομές. Αυτό είναι το πρώτο βήμα με περισσότερες πληροφορίες θα μπορούσαν να παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες σε άτομα ε, με ε, αναπηρίες παραδείγματο χάρη ώστε να γνωρίζουν αν προσφέρονται κάποια ειδικά βοηθήματα ε, στα μέσα μεταφοράς χρειάζεται δικτύωση αστικών μεταφορών ε, στο πλαίσιο των πολυτροπικών μεταφορών γιατί οι αστικές μεταφορές παρέχουν τη δυνατότητα ε, δικτύωσης ώστε να έχουμε μεταφορές από πόρτα σε πόρτα. Ακόμη δεν υπάρχει ε, κάτι που να εγγυάται τα δικαιώματα των επιβατών σε πολυτροπικές μεταφορές. Αυτό κάνει τις πολυτροπικές μεταφορές λιγότερο ελκυστικές. Πρέπει να φροντίσουμε να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα των πολυτροπικών μεταφορών γιατί αποτελούν καταρχήν το μέσο για να αποφύγουμε την υπερφόρτωση ε, των μέσων μεταφοράς που είναι τα περισσότερα εύκολα και θα παρέχουν και μεγαλύτερες δυνατότητες για τον τουρισμό στην Ευρώπη. Θα θέλαμε από την Επιτροπή τις γενικότερες διατάξεις που θα αποτελέσουν το πλαίσιο για καλύτερη ενημέρωση των επιβατών. Όσον αφορά τις υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων, η Επιτροπή θα πρέπει τον να αφήσει το θέμα αυτό στον ίδιο τον τομέα ώστε να αναζητηθούν οι κατάλληλες λύσεις δεν φαίνεται να υπάρχουν άμεσα κάποιες έτοιμες λύσεις, αλλά αν μέχρι το 2020 ο ίδιος το τομέας δεν καταλήξει σε λύσεις, θα μπορούσε να παρέμβει η Επιτροπή με δικές της προτάσεις. Οι πολυτροπικές μεταφορές είναι αυτές που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αποφύγουμε ε, προβλήματα και διαταραχές στις μεταφορές και ε, θα ήθελα να τονίσω ότι χρειαζόμαστε την υποστήριξη για να έχουμε καλύτερες προτάσεις στον τομέα των μεταφορών. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να προκύψουν από του ίδιου τους φορεί, από τον τομέα και από την Επιτροπή. Ελπίζω ότι θα έχω την υποστήριξή σας στην Ολομέλεια και ευχαριστώ εξ αρχή και τους συναδέλφου και ε, του βοηθού μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και αρχίζει η διαδικασία Κατσουδιάη με τον κύριο Φραντζούλητσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική η έκκληση προς τα κράτη-μέλη για κοινόχρονο διάγραμμα και ανταλλαγή πληροφοριών και επίσης ε, την ανάπτυξη υπηρεσιών εκδοσιστηρίων ε, για πολυτροπικές μεταφορές. Θα πρέπει να έχουμε πολυτροπικέ διασυνοριακές μεταφορές και αντίστοιχο σχεδιασμό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει την δημιουργία τέτοιου πολυτροπικού τρόπου έκδοση εταιρείων και αν δεν γίνει κάτι τέτοιο μέχρι το 2020 να αναλυθούν νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Μέσω στα χρονοδιαγράμματα και δίκαιη ανταλλαγή πληροφοριών, με ανοιχτέ διεπαφέ σε διαπεριφερειακό, εθνικό και κοινωτικό επίπεδο, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σχεδιασμό πολυτροπικών μεταφορών προ όφελο όλων των εμπλεκομένων. Σα ευχαριστώ κύριε Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αναβάθμιση των ευρωπαϊκών μεταφορών θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τον επιβάτη και όπως καταδεικνύει και η έκθεση, η σωστή παροχή έγκυρων πληροφοριών αποτελούν το πρώτο βήμα προς την πορεία αυτή. Για να καταφέρουν όμως να αναπτυχθούν οι πολυτροπικές μετακινήσεις τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και του τουρισμού θα πρέπει να τις καταστήσουμε πιο ανταγωνιστικές όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών το σύστημα κρατήσεων και αγορών στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι πιο απλό και διαχειρίσιμο από όλες τις ηλικίες και ιδίως από τους ηλικιωμένους. επίσης θα πρέπει να προβλέπονται μειωμένες τιμές για τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους και να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στις ειδικές τους απαιτήσεις όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού το σύστημα κρατήσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ευρωπαϊκής ένωσης και να προβλέπονται μειωμένες τιμές για φοιτητές ανέργους και πολύτεκνες οικογένειες. τέλος το εισιτήριο πολυτροπικών μετακινήσεων θα μπορούσε να ενταχθεί στα τουριστικά πακέτα διακοπών με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη προσέλκυση τουριστών. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Επίτροπε Μπούλτσα, ε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ καταρχήν τον κύριο Κόχ για την ε, εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για την έκθεση του. Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι υπέρ της ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εταιρείων. Καταρχήν, χρήση τις σύγχρονες τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας ε, στον τρόπο ε, κράτησης και αγοράς εισιτηρίων ε, για πολυτροφικές μεταφορές. Ε, για να αποφευθεί επίσης αθέμητος ανταγωνισμός. Και με τη χρήση νέων, νέων τεχνολογιών θα δημιουργήσουμε περισσότερες, πιο, πιο αποτελεσματικό σύστημα, θα μειώσουμε και τον αντίκτυπο προς το περιβάλλον, θα μειώσουμε τις ενεργειακές τιμές. Επίσης, θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών, γιατί ε, με, τη, με τη διευκόλυνση των μεταφορών προσπίζουμε τη βασική ελευθερία της διακίνησης των προσώπων. Ο κύριος αναφέρεται και η συγκεκριμένη επιλογή της ε, ε, μετακίνησης με ταχύ. Αυτό δεν είναι επιλογή, είναι περισσότερο αναγκαιότητα. Εγώ για να πάω από το σπίτι στο γραφείο μου ε, θέλω 35 λεπτά με το αυτοκίνητο και 4-5 ώρες με τις ε, αστικές συγκοινωνίες ε, και σκεφτείτε ότι πρέπει να επιστρέψω κιόλα. Δεν είναι θέμα λοιπόν επιλογή μόνο η χρήση του γιοταχή. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τι μαζικέ μεταφορέ πολύ πιο αποτελεσματικέ. Να μην έχουμε μόνο τα αντικίνητα αλλά και τα κίνητρα. Επίση, είναι οι πολυτροπικέ μεταφορέ βολικέ για όσου έχουν κοινά χερσαία σύνορα ή για τους μετακινούμενους διασυνοριακά. Αυτοί θα βοηθηθούν ιδιαίτερα, αλλά μην ξεχνάτε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι νησί ουσιαστικά. Οπότε το διοικητικό κόστος ενός τέτοιου καθεστώτος και το κόστος της εναρμόνισης κατά πάσα πιθανότητα θα υπερβεί το όφελος που θα αποκομίσει το Ηνωμένο Βασίλειο από ένα τέτοιο σύστημα. Ο κύριος Ιάκοφτσης. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο σας και σας ευχαριστώ που ήρθατε τόσο αργά για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό για μας η παρουσία σας. Είναι πολύ σημαντική για μας η παρουσία σας, γιατί αυτό δίνει το εχέγγυο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φροντίσει για την θέσπιση ενός ε, ε, μια ολοκληρωμένη πολυτροπική έκδοση εταιρείων και κράτηση ε, εισιτηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα αποβεί ιδιαίτερα ωφέλιμο για τον τουρισμό, που είναι σημαντικός κλάδος οικονομικός για πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση, ιδιαίτερα για τις χώρες του Νότου. Και ακριβώς στον τομέα αυτό ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε ένα αξιόλογο έργο για να καταστήσουμε τον τουρισμό μας ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε μία δίκαιη ε, πρόσβαση της, στις τιμές των εισιτηρίων και αυτό χάρη στο διαδικτυακό κόσμο είναι πολύ πιο εύκολο. Ε, ανοιχτή λοιπόν ε, και θεμητή προσέγγιση και ανταλλαγή των πρακτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έστω και αργά χαιρόμαστε ιδιαίτερα κύριε, Επίτροπε που ήρθατε στην, στο Κοινοβούλιο και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο βουλευτέ. Η Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κύριο Κόχαλα και τα μέλη τη Επιτροπή των Μεταφορών, γιατί ήταν πολύ αξιόλογη αυτή η έκθεσή του, γιατί τονίζεται πόσο σημαντική είναι αυτή η ενημέρωση, η πληροφορία για τις πολυτροπικές μετακινήσεις για όλους τους Ευρωπαίους παντού. Και οπότε συμφωνώ που τονίζεται το γιατί τι γίνεται με τον τελικό χρήστη και τι γίνεται με το πόσο ωφελείται η κοινωνία. Ακριβώς ε, αυτό είναι το πνεύμα της ενιαίας ψηφικής αγοράς όπως την έχουμε προτείνει. Και οπότε πιστεύουμε ότι έτσι θα πετύχουμε τους στόχους μας να μειωθεί η βλάβη στο περιβάλλον, περισσότερη ασφάλεια και έτσι θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι μεταφορές. Θα έχουμε θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη για να τα καταφέρουμε. Θα πρέπει να είμαστε συμβατοί με τις ανάγκες της κοινωνίας και κυρίως ε, με τις ανάγκες των πόλεων. Θα πρέπει να έχουμε πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες και να έχουμε καλύτερη ενσωμάτωση, ολοκλήρωση των ε, πολυτροπικών μετακινήσεων και έτσι να έχουμε μια διαχείριση πιο αποτελεσματική και αυτό να αφορά και τις ε, μετακινήσεις ε, ανθρώπων αλλά και φορτίων. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, έτσι θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε ακριβείς πληροφορίες ως τον τελικό χρήστη. Ο στόχος είναι να έχουμε ένα τέτοιο πλαίσιο και ιδίω όσον αφορά την έκδοση εισιτηρίων, κάτι που μας έχει απασχολήσει και έχουμε προβεί σε κάποιες πρωτοβουλίες, αξιόπιστες πληροφορίες ε, για κάθε επιλογή ταξιδιού που υπάρχει και να γίνεται παρουσίαση χωρίς ε, διαφήμιση αλλά αντικειμενικά ανάλογα με τις γεωγραφικές ανάγκες, του γεωγραφικού εντοπισμό του κάθε χρήστη και να μην έχουμε τον ανταγωνισμό όσον αφορά ε, τα δεδομένα θα έχουμε εφαρμογή νομοθεσία στα κράτη-μέλη αλλά όσον αφορά τις πληροφορίες για τα ταξίδια θα πρέπει να δούμε πώς αυτά τα δεδομένα θα είναι πολυτροπικού χαρακτήρα. Αυτό δεν το έχουν πετύχει ακόμα. Τα δρομολόγια, όπως είπε το Κοινοβούλιο, για όλες τις ε, τους που να ε, υπάρχουν και έχουμε έτσι ευκαιρία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε για πρόσβαση στα δεδομένα και αυτό είναι θέμα διαφόρων πρωτοβουλειών και εξορισμού αυτό είναι η βάση για να έχουμε καλύτερο σύστημα, καλύτερες υπηρεσίες. Πολύ σημαντικό για να έχουμε ε, θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων. Πάρα πολύ σωστά το Συμβουλίο είπε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα των εισιτηρίων και διασυνοριακά και επίσης έχουμε κάποιες κρατικές πρωτοβουλίες τόσο ώστε οι μέτοχοι να βελτιώσουν τις συνθήκες όπως επίσης τα ευφύ εισιτήρια και τις συνδρομικές υπηρεσίες. Συμφωνούμε 100% με το Κοινοβούλιο όσον αφορά το ότι θα πρέπει οι πληροφορίες να είναι συμβατές με τις ανάγκες όλων, ακόμα και των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας. Να έχουμε στην αγορά ε, διαφάνεια και να μην υπάρχουν δυσμενείς διακρίσεις και να είναι καλά περιχαρακωμένα τα δικαιώματα των χρηστών, ιδιωτικότητα, οπότε έτσι να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες και τέλος τα δικαιώματα των επιβατών για τις πολυτροπικές μετακινήσεις. Εμείς τώρα ασχολούμαστε με αυτό και θα κάνουμε μια έκθεση επιπτώσεων όσον αφορά τις διαφορετικές εναλλακτικές, ώστε όλοι οι επιβάτες να έχουν κατοχυρωμένα τα δικαιώματά τους. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε.